Όχι. Η κυρία Λένα Κολάρσκα Μπομπίνσκα ε, ανέλαβε ε, Υπουργός ε, Πολιτικής Επιστημών και ο κύριος Ράφαλ Τρασκόφσκι ε, ανέλαβε το Υπουργείο Διοίκησης και Ψηφιακού Θεματολογίου του συγχαίρουμε. Ε, χειρεύουν οι θέσεις από 3 Δεκεμβρίου και ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Η Νομική Επιτροπή ε,